θα γίνει αύριο. Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η προφορική ερώτηση που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μογγολία. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχήν στο συντάκτη μας, στον κύριο Μπαρτολότσι, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η αντιπροσωπεία για τη σχέση με την Κεντρική Ευρώπη και Ασία είχε την ευκαιρία να μεταβεί στη Μογγολία μερικές εβδομάδες πριν. Ήταν πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα εμπειρία. Η Μογγολία είναι μια χώρα την οποία θα πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα και δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες να τις προσδώσουμε τη σημασία που της αρμόζει. Πρόκειται για μια χώρα που έχει ένα πολιτικό σύστημα συμμετοχής πολλών πολιτικών κομμάτων, δηλαδή ένα πλουραλιστικό σύστημα και τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα πολύ καλύτερα από άλλες χώρες της περιοχής εκείνης. Σε σχέση με το θέμα του περιβάλλοντος υπάρχουν δυσκολίες διότι υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη απερίμωση. Παράλληλα πρόκειται για μια χώρα η οποία έχει μεγάλο φυσικό πλούτο, ουράνιο, χαλκό, λευκοσίδηρο, άνθρακα και άλλα. Για αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη Μογγολία σε αυτή την κρίσιμη φάση της ανάπτυξής σας και να μιλήσουμε για την ενίσχυση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν οι φυσικοί πόροι της χώρας για την ευημερία των πολιτών της. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε τη Μογγολία στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να φτάσει στα δικά μας επίπεδα μιας οικονομίας της αγοράς και μιας καλής βιομηχανίας. Θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου στη χώρα αυτή και τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα στα πλαίσια αυτά η Συμφωνία Οικονομικών Εταιρικών Σχέσεων θα πρέπει να ενισχυθεί μαζί με 45 συναδέλφους υποβάλαμε αυτή την προφορική ερώτηση ζητώντας περισσότερες πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας και τις δυνατότητες, μάλλον και του χρονοδιαγράμματος κύρωσης της συμφωνίας. Η μονογραφή έχει ήδη γίνει, αλλά όχι η τελική υπογραφή. Επειδή μία χώρα εκφράζει αμφιβολίες ως προς την νομική βάση που χρησιμοποιείται. Επίσης θα θέλαμε να ρωτήσουμε την Επιτροπή για το τι δυνατότητες υπάρχουν για να ανοίξουμε ένα γραφείο στην πρωτεύουσα της Μογγολίας και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την οικονομική και πολιτική συνεργασία με τη χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Φίλε εξ της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής θα ακούσει με μεγάλη χαρά φαντάζομαι τις τελευταίες εξελίξεις που συζητιούνται για τη σχέση μας με τη Μογγολία. Είναι η 19η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου και βρίσκεται σε στρατηγικό σταυροδρόμι αναπτυσσομένων αγορών μεταξύ Ρωσίας και Κίνας είναι χώρα με μακρά και λαμπρά παράδοση και έχει επιλέξει το δρόμο της δημοκρατίας. Την συγχαίρω για τις ειρηνικές εκλογές που διεξήχθησαν εκεί πρόσφατα. Είναι ένα ακόμα βήμα προς τον δρόμο της Μογγολίας, προς τον πολιτικό πλουραλισμό. Εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το μορατόριο επί της θανατικής ποινής που επιβάλλει πλέον η Μογγολία και όπως το ζήτησε και εκείνη είμαστε έτοιμοι να της διαθέσουμε τεχνογνωσία για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών και προτύπων. Χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να πω ότι η Μογγολία συμπεριλαμβάνεται στις πιλωτικές χώρες στήριξης της δημοκρατίας από την Ένωση. Θα τις δώσουμε δηλαδή μια μικρή χρηματική και τεχνική βοήθεια. Επίσης με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να τη συγχαρώ για την ε, εκατονταετή επέτειο που γιόρτασε φέτος της κρατικής της υπόστασης. <clears throat> για την οικονομική της ανάπτυξη θα έλεγα τα εξή. Βρίσκεται και οικονομικά σε σταυροδρόμι γιατί από βουκολική κοινωνία και νομαδική γίνεται σύγχρονη οικονομία. Έχει διαθέτει τεράστιο ορυκτό πλούτο που είναι μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα αυτή για να δημιουργήσει μεγαλύτερη ευημερία για το λαό της. Ελπίζουμε ο ανεκμετάλλευτος αυτός ο ρηκτός πλούτος να αποτελέσει ευλογία μάλλον παρά κατάρα για τη χώρα όπως έγινε για άλλες ορισμένες περιπτώσεις σε άλλες χώρες. Για τις διεθνείς σχέσεις εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή της σε αποστολές του ΟΗΕ για την ειρήνευση διαφόρων περιοχών του κόσμου μαζί με το Κονγκό, ε, στο Κονγκό του Σουδάν, την Δυτική Σαχάρα του Τσάντα. Ναι. Και θα ήθελα να τονίσω ότι οι προσπάθειες της Μογγολίας για τη σταθεροποίηση του Αφγανιστάν είναι επίσης κάτι που εκτιμούμε ιδιαίτερα. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση και τις σχέσεις της Μογγολίας με την Ένωση, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η συμφωνία συνεργασίας που αντικαθιστά την προηγούμενη έχει τύχει διαπραγμάτευσης και εγκριθεί από τις 20 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους στην Ουλάν Μπατόρ. Η συμφωνία αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας. Είπατε εκπρόσωπος ε, και αντιπρόεδρος η κυρία Άστον καλωσόρισε τη συμφωνία αυτή ως και αναφέρω κατά λέξη άλλο ένα βήμα προς την ενισχυμένη οικονομική και πολιτική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της με τη Μογγολία. Με την συμφωνία αυτή θα συνεργαστούμε ως ισότιμοι εταίροι σε μια σειρά θεμάτων από πολιτικά ζητήματα όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέχρι το εμπόριο και τις επενδύσεις σε τομείς σημαντικούς όπως οι πρώτες ύλες. Μόλις εγκριθεί το κείμενο από τα κράτη-μέλη, ελπίζουμε να μπορέσουμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό για να έρθει στις Βρυξέλλες να υπογράψει την συμφωνία με την ύπατη εκπρόσωπο. Δεδομένης της εμβάθυνσης της συνεργασίας μας και της ε, θέσης σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας ε, υπάρχει επιλογή του να ανοίξουμε μία αντιπροσωπεία της Ένωσης ε, στο Ουλάν Μπατόρ. Ελπίζω να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε οι οικονομικές δυσκολίες και δυσκολίες στον τομέα του προσωπικού για να ανοίξει μια πλήρης αντιπροσωπεία στην Ουλάν Μπατόρ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω τα σχολεία σας. Ευχαριστούμε. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Μικολάσης από το ΕΛΚ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Φίλε, συνάδελφοι, η σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μογγολίας την τελευταία εικοσαετία εξελίσσονται θετικά. Και αυτό είναι απότοκο του εκδημοκρατισμού και του εξυγχρονισμού στη Μογγολία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη για το μακροχρόνιο δημοκρατικό καθεστώς της Μογγολίας. Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να αναθεωρηθεί το δικαιοδοτικό σύστημα και να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Επίσης, θα πρέπει να κινηθεί η χώρα προς μια οικονομία της αγοράς με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις στον, στο τομέα του εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Πιστεύουμε ότι η χώρα Βλέπει την νομοθεσία έτσι ώστε να μην γίνεται ε, κακοχρησία της δεσπόζουσας θέσης ορισμένων επιχειρήσεων και την πρόθεση των καρτέλ. Είμαι πεπισμένος ότι έτσι θα ενθαρρυνθούν οι ξένοι επενδυτές και θα επενδύσουν σε αυτή τη χώρα στον, ε, στις περιφέρειες, στις αγροτικές περιφέρειες, οι πολίτες εξαρτώνται από την αγροτική οικονομία. Νομίζω ότι ο Επίτροπος Φιλ μίλησε για μία μόνιμη αντιπροσωπεία στη Μογγολία Πιστεύω ότι μπορούμε να προωθήσουμε τις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις γνωρίζοντας ότι, πρόκειται, ότι η Μογγολία διαθέτει μεγάλο ε, πλούτο, μεταλλευτικό πλούτο, μεγάλο ορυκτό πλούτο. Γι' αυτό νομίζω ότι οι σχέσεις μας θα πρέπει να ενισχυθούν. Ευχαριστώ, κυρία Ογιουλάντ από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Μογγολία έχει πολλές πρώτες ύλες, χαλκό, βουλφράμιο, λευκοσίδρο, χρυσό και άρα αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο, αλλά ταυτόχρονα βεβαίως θα πρέπει επί τη ευκαιρία και εμείς να επιβάλλουμε όρους για να ενθαρρύνουμε τη Μογγολία να ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη Μογγολία με καλπάζουσα διαφθορά, έλλειψη καλής διακυβέρνησης ε, και ελληματική διεθνή συνεργασία. Επιπλέον υπάρχουν κάποια ζητήματα με τη διαχείριση φυσικών πόρων αυτή τη στιγμή. Τα αποθέματα της Μογγολίας θα εκμεταλλεύονται πολλές ξένες εταιρείε με συνεργό την μογγολική κυβέρνηση. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία ο λαός της Μογγολίας δεν υποφελείται από τους πόρους της χώρας. Πρέπει, παραδείγματο χάρη, να εργάζονται στα ορυχεία με άθλιες συνθήκες, ε, κάνοντας εξόριξη με υδράργυρο που βλάπτει την υγεία και πολλά παιδιά γεννιούνται στη Μογγολία με ανίατες ασθένειες και παραμορφώσεις. Η οικονομία της Μογγολίας επίσης αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω και ε, δασμών και απαγορεύσεων εισαγωγών που τις επιβάλλουν η Κίνα και η Ρωσία αλλά και λόγω τεχνικών ελλείψεων. Η κτηνοτροφία αποτελεί γύρω στο 80% της αγροτικής παραγωγής αλλά το κρέας δεν μπορεί να εξαχθεί καλώς δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ποιοτικού ελέγχου. Εάν έχουμε στόχο ε, μια τέτοια συμφωνία, τότε πρέπει να βοηθήσουμε τη Μογγολία να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα για να απτυχθεί κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ από τους μη εγγεγραμμένους ο κύριος Κόβατς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πριν από τρεις εβδομάδες πήγα στην 8η αντιπροσωπεία στην Ουλάν Μπατόρ και είδα εκεί με τα μάτια μου ότι οι πολιτικές δομές και διευθετήσεις προχωρούν προς τον εκδημοκρατισμό. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επίσης σημειωθεί τεράστιες πρόοδοι και συναντήσαμε και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που μας εξήγησαν ότι είναι αναγνωρισμένες από την κυβέρνηση. Επίσης πρέπει να χαιρετήσουμε την ελευθεροτυπία που βασιλεύει εκεί. Με αυτή τη συμφωνία συνεργασίας έχουμε μπροστά μας ένα ακόμη βήμα μέσω του οποίου να χορηγήσουμε τεχνογνωσία στη Μογγολία. Το γραφείο εκπροσώπησής μας εκεί είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να βελτιωθούν οι σχέσεις μας. Τώρα είμαι μονομένοι ομιλητέ. ο κύριος Ζέλερ πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπαρτολότσι που έλαβε την πρωτοβουλία και έκανε θέμα συζήτηση στη Μογγολία. Ξέρετε πώς αντιμετωπίζουμε διαφορετικά το κάθε πρώην Σοβιετικό κράτος η δε Μογγολία παραμελήθηκε και αυτό είναι άδικο γιατί χρησιμοποίησε νωρί την ανεξαρτησία της και εκδημοκρατίστηκε η Μογγολία. Ήδη το 1992 είχαν δημοκρατικό σύνταγμα, έκτοτε έχουν λάβει χώρα πολλές εκλογές ε, και όλοι οι παρατηρητές συμφώνησαν πως ήταν δημοκρατικές, κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο για τα κράτη εκείνης περιοχή. περιοχής. Η μογγολική κυβέρνηση προσπαθεί εδώ και κάποια χρόνια να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Το 2010 επέβαλε ένα μορατόριουμ για τη θανατική ποινή, κάτι που δεν έχουν κάνει άλλες δημοκρατικές χώρες. Βεβαίω τα 3 εκατομμύρια αυτή τη τεράστια ε, χώρα ε, με τα ακραία ε, κλιματικά φαινόμενα εξακολουθούν να ζουν μια νομαδική ζωή και υπάρχουν λίγες πόλεις που δεν έχουν ε, υποδομές. Ήδη εκμεταλλεύονται το υπέδαφος της χώρας, υπάρχουν κάποια ενεργειακά προβλήματα και η χώρα είναι στριμωγμένη μεταξύ Ρωσίας και Κίνας και εξαρτάται από αυτές τις χώρες. Βεβαίως θα πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε τον εκδημοκρατισμό, ο οποίος είναι υποδειγματικός για εκείνη την περιοχή του κόσμου. Και η ε, Μογγολία θα πρέπει βεβαίως ε, να έχει και άμεση εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρωτεύουσά για να δείξουμε πως δεν μας είναι διάφοροι. Μία πρόταση ακόμα, δώστε μου. Λυπούμε για το ότι δεν ήταν διατεθειμένη η διάσκεψη των Προέδρων να μας επιτρέψει και ένα ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ρινάλντι για ένα λεπτό. Σε σχέση με το άνοιγμα της αντιπροσωπείας του Λαμπατόρ που θα πρέπει να δοθή σε αντιπαράθεση με τη θέση του Πεκίνου. Γνωρίζουμε όλοι ότι η χώρα έχει μεγάλο ορυκτό πλούτο, αλλά υπάρχουν πολλές μορφές κοινωνικής αδικίας. Θα ήθελα η Επιτροπή να μας πει πώς, ε, θέτει, πώς λαμβάνει υπόψη τη Μογγολία ως προς την γεωστρατηγική της θέση. Ίσως θα μπορούσαμε να προβάλλουμε μία στρατηγική όπως ισχύει για τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και όπως την έχει εκπονήσει η Επιτροπή. Πρόκειται για μία χώρα παρατηρητή στον ΟΑΣΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται να βοηθήσει τη Μογγολία για να γίνει πλήρες μέλος του ΟΑΣΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους, πολι... τους πολιτισμικούς δεσμούς Μογγολίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Μπασέσκου. Κύριε Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να ε, συγχαρώ τον κύριο Μπαρτολότσι για αυτή τη ε, πρωτοβουλία. Οι σχέσεις Μογγολίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ειδωθούν υπό την οπτική γωνία της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Έτσι θα ενθαρρυνθεί η οικονομική συνεργασία. Η Μογγολία έχει ε, μεγάλο ενεργειακό δυναμικό και αποθέματα οι σχέσεις μας βασίστηκαν μέχρι δε στις εμπορικές σχέσεις μετά το 1993. Έκτοτε δεν είχαμε πολλές και ενισχυμένες εμπορικές σχέσεις. Έγιναν ανταλλαγές φοιτητών και πιστεύω ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε το πρόγραμμα Εράσμους μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας. Χρειάζεται μία αντιπροσωπεία μας εκεί για, την, για τον καλύτερο συντονισμό αυτών των δραστηριοτήτων. Έτσι οι επαφές με τις αρχές θα μας βοηθήσουν μέσα στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ως γνωστόν πλούσια σε πετρώματα και οι κινέζικες εταιρείες έχουν πάρει δικαιώματα εκμετάλλευσης και ασκούμε κριτική στις ε, κινέζικες εταιρείες για το ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό στην εξόριξη και εξεραίνουν τη στέπα. Επίσης υπάρχουν και οι διαμαρτυρίες των ε, Μογγόλων και ξέρετε πως είχαμε Άρα άλλο ένα ανοιχτό θέμα πέρα από τους Ουιγούρους ε, και τους Τιβετιανούς για την Κίνα. Και από ό,τι φαίνεται θα ενταθεί αυτή η σύγκριση. Οπότε πλέον αυτό το θέμα αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα και στη Μογγολία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη για την θετική του συνεισφορά για το θέμα της Μογγολίας. Σύντομη η συζήτηση, αλλά άκρο ενδιαφέρουσα για αυτόν τον εταίρο που αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερόμενο σε ένα ή δύο ζητήματα που εθίγησαν κατά την συζήτηση, θα ήθελα να πω, Πρόεδρε, ότι η Συμφωνία Εταιρικής ε, Σχέσης και Συνεργασίας, Οικονομικής Συνεργασίας, καλύπτει τις, τα βασικά πρότυπα και προδιαγραφές, βιώσιμη ανάπτυξη, περιλαμβάνοντας το περιβάλλον και το κοινωνικό περιβάλλον, ε, τρίτον εμπόριο και πρώτες ύλες, και την δικαιοσύνη, της ελευθερίας, καθώς και το θέμα της μετανάστευσης. Ως προς το χρονοδιάγραμμα, το κείμενο έχει υποβληθεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να υπογράψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Βουλή των Κοινοτήτων, γίνεται εξέταση του θέματος σε σχέση με το opt και σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Εξ ονόματος της ε, Βουλής των Αντιπροσώπων, μάλλον θα ήθελα να πω ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ενδεχομένως η υπογραφή, η τελική υπογραφή να γίνει το Σεπτέμβριο στην επόμενη συνεδρίαση της κοινή Επιτροπής Μογγολίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και μας χωρίζουν οι μεγάλες αποστάσεις, μεγάλη απόσταση, η αρρωγή μας είναι μεγάλη, υπάρχει ανοιχτό πνεύμα στη ε, Μογγολία και μεγάλη ανεκτικότητα ως προς τα πλαίσια του ΣΟΕΣ. Θεωρούμε ότι είναι η τρίτη γείτονα χώρα, όχι μόνο στα λόγια και στις ε, πράξεις. Και τέλος, θα ήθελα να επανέλθω ένα άλλο θέμα το οποίο ξέχασα σε σχέση με τον ΟΑΣΕ. Θα γίνει μια ειδική συνάντηση αύριο στη Βιέννη μέσα στα πλαίσια του Μονίμου Συμβουλίου του ΟΑΣΕ. Τα κράτη-μέλη θα ακούσουν τον Υπουργό Εμπορίου, Εξωτερικού Εμπορίου της Μογγολίας και μπροστά μου έχω τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να σας πω ότι θα τονίσω ότι προσβλέπουμε στη συνεργασία μας και μέσα στα πλαίσια του ΟΑΣΕ και τη συνεργασία της ε, Μογγολίας. Και επειδή η Μογγολία προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ε, δεσμεύσεις, έχει τη δυνατότητα να είναι ένας πολύ καλός συνεταίρος σε αυτή την περιοχή. Η συζήτηση έχει λήξει. Έχω μία ανακοίνωση, έλαβα από την ομάδα μεταρρυθμιστών, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών έναν κατάλογο διορισμών που θα ενταχθούν στα, πρακτικά εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς τους διορισμούς αυτούς. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει αύριο 5η 9 του μήνα.